φορικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τίτλος της οδηγίας θα ανακοινωθεί στα πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης. Θα υπάρξει ένα διάστημα τριών μηνών για να ε, εκφράσει την άποψή του το Κοινοβούλιο η οποία ξεκινά από αύριο στις 10 Ιουνίου 2016. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη λοιπόν σήμερα το απόγευμα είναι η προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν